τους συναδέλφους που άκουσαν και τους άλλους ε, συναδέλφους να ευχαριστήσω τον, τον Επίτροπο Ντάλη που έμεινε μέχρι τόσο αργά. Ολοκληρώνεται λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση. Επόμενη